τον αριθμό των ψηφιζάντων αλλά και των όσων ψήφισαν υπέρ ή κατά. Θέλαμε να απλοποιήσουμε τα... Ε, η ζωή μας, αλλά ε, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ψηφίζουμε την έκθεση Κοέλιο για τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και των βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έχει αποσυρθεί τροπορφορική τροπολογία και ψηφίζουμε την τροπολογία 1 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία, το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 594 ψήφους υπέρ, 51 ή κατά 37 αποχές. Προχωράμε τώρα, συγχαρτήρια καταρχήν στον εισηγητή. Ο κύριος Περώνη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ε, διάταξη των εργασιών. Είπατε ότι μετά από αίτημα των δημοσιογράφων, ε, μια καθόλου αξιοσεβαστή κατηγορία, θα ανακοινώνεται όλες τις ψηφοφορίες. Όμως νομίζω ότι ε, ψηφίζουν οι βουλευτές και όχι οι δημοσιογράφοι. Αυτός ο σύνδεσμος των δημοσιογράφων είναι των τυφλών. Είναι σύνδεσμος τυφλών δημοσιογράφων. Διότι οι δημοσιογράφοι μπορούν κάλλιστα να βλέπουν στις οθόνες την έκβαση της ψηφοφορίας κάθε φορά. ίσως σηκωθεί να έχουν μετά πρόβλημα οι δημοσιογράφοι, αν εσείς απλώς λέτε τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε κύριε Σπερώνη, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω προσωπική κρίση για τις δυσκολίες ε, της εργασίας των δημοσιογράφων. Όμως αυτό το αίτημα έφτασε στο Προεδρείο αυτή τη στιγμή, άρα θεωρώ ότι και προσωπικά συμμερίζομαι τη δική σας, ε, το δικό σας προσανατολισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει την απάντηση θα πρέπει να τη δώσει το Προεδρείο και προβλέπεται ήδη ε, για την ημερήσια διάταξη του επόμενου Προεδρείου ε, η υπόθεση αυτή. Παρακαλώ, ο κύριος Μακμίλαν Σκότ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τη θέση του κυρίου Σπερώνη. Αναγνωρίζω τη δυσκολία στην οποία βρίσκεστε εσείς, αλλά νομίζω πως έχει δίκιο. Γιατί στις οθόνες όντως καταγράφονται όλες οι ψήφοι, όμως το να διαβάζουμε, διαβάζετε κάθε φορά αποτελέσματα είναι πολύ χρονοβόρο, ιδιαίτερα ε, για ε, τη δουλειά που έχουμε. Εγώ προτείνω να παραπέμψετε το θέμα στην αρμόδια επιτροπή, αν το δέχεται και το σώμα. Όπως είχα ήδη πει, το Προεδρείο θα αναλάβει να εξετάσει το θέμα, ακριβώ για να δώσει οριστική απάντηση. Λοιπόν, η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψήφιση τη έκθεση του κυρίου Λάμστορφ για το συντονισμό των διαδικασιών ε, στους δημόσιους ομοιοδοτικούς διαγωνισμούς για έργα, εξοπλισμού ή υπηρεσίες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Ποιοι είναι υπέρ της πρώτης συμβαστικής. Ευχαριστώ. Το πρώτο, η πρώτη δέσμη συμβαστικών ε, εγκρίνεται και καταπίπτει το δεύτερο, η δεύτερη δέσμη. Η πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομαστική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 597 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημα, μπορεί να έρθει κάποιος τεχνικός. Αλλά 299. Ordine del giorno, votazione sulla relazione. Λοιπόν, έκθεση Σλάιτερ. Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα. Και εδώ έχουμε ε, μια, πρώτη δέσμη, συμβιβαστικές τροπολογίες, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά η δεύτερη δέσμη, ψηφίζουμε για την τροποποιημένη πρόταση υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Απροβάτα τη Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 674 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Προχωράμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Φιγκερέντο για την εξουσιοδότηση κύρωση τη Σύμβαση τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα τη αλληλεία του Διεθνούς Οργανισμού, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε άρχεται ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 671 ψήφους υπέρ. Συγχαρτήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση Κατάνια για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2004 με 2008. Ψηφίζουμε για το αρχικό κείμενο της παραγράφου υπαριθμών 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 3. Προχωράμε στην τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 17 είναι μια ψηφοφορία σε χωριστά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, πρέπει να επαληθεύσουμε. Οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 346 ψήφοι υπέρ, 332 κάτα, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 18 σε χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Ορίστε ψηφοφόρια για την παράγραφο 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προχωράμε τώρα στην ψηφοφορία για την παράγραφο 23. Αρχικό κείμενο, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος Α, όχι. Τροπολογία 32 ε, στην παράγραφο 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως... Αλλά ας το επαληθεύσουμε καλύτερα. Λοιπόν, για την τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία με 382 ψήφους ε, υπέρ και 303 κατά. Προχωράμε τώρα στην τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για την παράγραφο 30 τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία του αρχικού κειμένου με πέντε χωριστά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά Ας επαληθεύσουμε για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα της παραγράφου 30. Τέλος της ψηφοφορίας. 433 υπέρ. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και το πέμπτο τμήμα. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για την παράγραφο 31 έχουμε χωριστή ψηφοφορία για δύο τμήματα με ονομαστική ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 521 ψήφους. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 598 ψήφους υπέρ. Εγκρίνεται ολόκληρο παράγραφο δηλαδή. Πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχουμε λοιπόν για την παράγραφο 32 ψηφοφορία σε τμήματα για το αρχικό τμήμα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπάρχει έτοιμα προφορικής τροπολογίας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι για να συμπληρώσω το κείμενο αυτής της τροπολογίας που Θέλω να προσθέσω μετά από το κείμενο που λέει 12 Δεκεμβρίου 2006 να προσθέσουμε και στις 4 και 17 Δεκεμβρίου 2008. Γιατί ελήφθησαν αποφάσεις από το δικαστήριο σε αυτές τις ημερομηνίες και δεν θα ήταν σωστό να αναφέρουμε την απόφαση του 2006 χωρίς αναφέρουμε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν το Δεκέμβριο του 2008. Το καταλάβατε όλοι, ελπίζω. Θα μπει στο πρώτο τμήμα του κειμένου που ψηφίζουμε. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Οπότε ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. υπέρ κατά αποχές νομίζω πως απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία La votazione Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 368 ψήφους κατά έναντι 237 υπέρ. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα με χωριστή πάλι ψηφοφορία κατά τμήματα την παράγραφο υπαριθμών 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 25. Με αναφερά στο τμήμα Β. Στο σημείο Β, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τον κατάλογο ψηφοφοριών, φαίνεται ότι η παράγραφος 36 έχει προσυρθεί. Έπρεπε να την ψηφίσουμε ή όχι. Ε, ναι, έχει αποσυρθεί η τροπολογία 8 και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για την παράγραφο 36. Ας επανέλθουμε λοιπόν στην ψηφοφορία της τροπολογίας 25 που σχετίζεται με την παράγραφο 38 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 366 κατά 299 υπέρ. Τροπολογία υπερθμός 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα δεν έχετε μετάφραση. Δεν υπάρχει μετάφραση. Α, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να αλλάξω γλώσσα γιατί ούτω ή άλλω θα μεταφράζεται και τα αγγλικά αν μιλάω αγγλικά. Πάμε στην παράγραφο 45. Ψηφίζουμε για το αρχικό κείμενο υπέρ. Ποιο είναι το πρόβλημά σα. Α, προσπαθώ να σας ερμηνεύσω για την παράγραφο 40. Αφού εγκρίναμε την τροπολογία υπαριθμών 43, καταπίπτει η ψηφοφορία για ολόκληρη την παράγραφο και άρα και η ψηφοφορία για το... με χωριστή, ψηφοφορία σε τμήματα. Λοιπόν, άρα πάμε στην παράγραφο 45. Υπέρ, ποιοι είναι παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 10. Συγγνώμη, 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα πάμε... Α, θέλετε να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Τροπολογία 35 για την παράγραφο 49. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. 452 υπέρ, 211 κατά. Εγκρινέται. Παράγραφος 51. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο σε πέντε διαφορετικά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 619 ψήφους. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 344 ψήφους υπέρ. 323 κατά. Τρίτο τμήμα. Εγκρίνεται με 627 ψήφους. Τέταρτο τμήμα. Votazione chiusa. Approvato con 560. Τέλος της ψηφοφορίας. 569 ψήφοι υπέρ, εγκρίνεται. Τελευταίο τμήμα, ψηφίζουμε. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Και αυτό εγκρίνεται. 367 ψήφοι υπέρ. Άρα λοιπόν ολόκληρη παράγραφος 51 εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στην ψήφιση της ε, παραγράφου 55 τέταρτο εδάφιο του αρχικού κειμένου σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κοντράρια Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 25, 21 ε, συγγνώμη, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατά συνέπεια πάμε να ψηφίσουμε στο αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα και τα δύο με ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. 651 μία ψήφη υπέρ. Ε, δεύτερο τμήμα άρχεται ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Και αυτή εγκρίνεται με 427 ψήφους υπέρ. Και τώρα πάμε στη τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε στο αρχικό κείμενο της ε, παραγράφου 62 σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Τώρα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione Τέλος ψηφοφορίας. 407 υπέρ εγκρίνεται. Πάμε σε ψηφοφορία σε δύο τμήματα για την παράγραφο 65. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κείμενο της παραγράφου 71. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 29 με ονομαστική ψηφοφορία για την, τροπολογία, για την παράγραφο 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 367 ψήφους υπέρ. Πάμε τώρα στην παράγραφο... Μετά, μάλλον, από την παράγραφο 72, τροπολογία 30, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 591 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Τέλος. Τροπολογία 53 για την παράγραφο 73. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 73 ψηφίζουμε τώρα σε χωριστά τμήματα. Τι Θέλετε παλήθευση. Εντάξει. Παράγραφος 73, τροπολογία 53. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. 317 υπέρ, 353 κατά. Απορρίπτεται. Λοιπόν, τώρα το αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Περνάμε στην τροπολογία 54 για την παράγραφο 75. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται με 403 ψήφους κατά. Τροπολογία 22, παράγραφος 76, ονομαστική ψηφοφορία. La votazione è... Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 401 ψήφι υπέρ. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το κείμενο της παραγράφου 78 με χωριστά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται πως εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά Λοιπόν, ψηφίζουμε για την τροπολογία 36. La votazione è chiusa. Approva... Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 404 ψήφους, άρα καταπίπτει 58 και δεν ψηφίζουμε και για το αρχικό κείμενο. Πάμε στην τροπολογία 44, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε για την παράγραφο 90 στο αρχικό, στο αρχικό της κείμενο σε δύο χωριστά τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατά συνέπεια ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 92 σε τρία χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και το τρίτο τμήμα. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 100. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος ε, ε τροπολογία 45, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Ε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 296 ψήφοι υπέρ, 379 κατά. Άρα ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την αρχική παράγραφο υπαριθμών 103. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 396 ψήφοι υπέρ. Τώρα, παράγραφος 104. Εδώ, Ψηφίζουμε για το σύνολο του παραγράφου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 105 χωρίς τη ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 για την παράγραφο 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν για το αρχικό κείμενο της παραγράφου 107 σε 6 χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απο... Ε, εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έξτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπράβο, καλή γυμναστική κάνετε. Παράγραφος 108 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρο... Παράγραφος 111. Τροπολογία 39. Υπέρ. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Τώρα έχουμε φτάσει στην παράγραφο 120. Αρχικό κείμενο. Δύο χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε φτάσει, έχει φτάσει με μια μικρή γραφειοκρατική καθυστέρηση ένα αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Ακόμα και δεν υπάρχει στον κατάλογο των ψηφοφοριών, ε, α το δεχτούμε την ονομαστική ψηφοφορία. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν με ονομαστική ψηφοφορία την 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 531 ψήφοι κατά. Τροπολογία 60. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό τμήμα της παραγράφου 149. Δύο χωριστά τμήματα, με ονομαστική ψηφοφορία. Για το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε πρώτα. Τέλος της <laughs> ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 640 ψήφοι υπέρ. Δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Votazione chiusa. 330... 334 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Πάμε στο αρχικό κείμενο της 157. Δύο χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 για την παράγραφο 159 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο της 159 το αρχικό σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παρακαλώ. Παράγραφο 166. Για την 166 να σας πω ότι το αρχικό κείμενο στα αγγλικά είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε γιατί υπάρχουν διάφορες ε, μεταφράσεις που αλλάζουν τελείως τη μετάφραση η, ας πούμε, η, ακόμα και η Ιταλική εκδοχή είναι λάθος. Πάντως αυτό που ισχύει είναι το αγγλικό κείμενο. Σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε, θα το ψηφίσω, θα το θυμίσω κι εγώ, αλλά τώρα είμαστε ακόμα στην 161. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε και για το αρχικό κείμενο της 161, αφού απορρίψαμε την τροπολογία τη σχετική. Υπέρ λοιπόν, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 166. Να επαναλάβω ότι το σωστό κείμενο είναι το αγγλικό, γιατί υπάρχουν πολλά λάθη στη μετάφραση. Ψηφίζουμε λοιπόν την 166 με ονομαστική ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 374 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται το κείμενο. Και τώρα, να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφόρια το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. La votazione è chiusa. 400... Τέλος της ψηφοφορίας. 401 ψήφι υπέρ, έναντι 220 κατά. Εγκρίνεται το ψήφισμα συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία του ψηφίσματος της Επιτροπής ε, ε, Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη Σύμβαση για την Εργασία των Ναυτικών για το 2006. Η συγκίτρια είναι η κυρία Μακδόναλτ. Ψηφίζουμε τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία το ψήφισμα στο σύνολό του. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. 646 ψήφοι υπέρ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εγκρίνεται το ψήφισμά της. Και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Αντρικένε για την ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη δέσμη τροπολογιών από το 1 το 7 έχει υποβάλει η συγγήτρια υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψήφισμα στο σύνολό του. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, είπα. Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμα, αλλά εντό ολίγου θα έχει αρχίσει. Μια ρέντο. Παραδίδομαι. Α, να. Votazione chiusa. 629 voti favorevoli. Abbiamo... 629 ψήφοι υπέρ εγκρίνεται το ψήφισμα. Συγχαρτήρια. Και τώρα πάμε στην έκθεση του κυρίου Καπάτο για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Λοιπόν, δύο κομμάτια, δύο τμήματα χωριστά υπέρ του πρώτου τμήματος κατά ε, γκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφορία για την παράγραφο 4. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κείμενο της παραγράφου 5, η παύλα, σε έξι χωριστά τμήματα, υπέρ του πρώτου τμήματος, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Λοιπόν, έλεγχος για το τέταρτο τμήμα. Τέταρτο τμήμα της παραγράφου άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Τέλος. 374 υπέρ εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται και το δέκτο τμήμα. Άρα ολόκληρη παράγραφος. Πάμε τώρα. Πάλι. Παράγραφος 5. Τρίτη παύλα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Υπέρ, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11, παύλα 4, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Credo Scusate, forse ho fatto un errore, ma Ίσως έκανα λάθος, αλλά... Εν πάση περιπτώσει, θα επαληθεύσουμε. Παράγραφος 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Μόνο 176 υπέρ και 421 κατά. Όχι απλώς απορρίπτεται, αλλά απορρίπτεται τελείως. Καταπορρίπτεται. Υπεραπορρίπτεται. Λοιπόν, παράγραφος 20. εγκρίνεται. Παράγραφος 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο recital. στο εκτιμώντας F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του. Με ονομαστική ψηφοφορία, τέλος της, ε, άρχεται η ψηφοφορία, με συγχωρείτε. La votazione 355 voti. Τέλος ψηφοφορίας, 355 υπέρ, 195 κατά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τέλος των ψηφοφοριών. Και ενώ εγκαταλείπετε την αίθουσα, θα αρχίσουμε με τις δηλώσεις επεξηγήσεις ψήφου. Allora, relazione Coelho. Έκθεση Coelho. Mr. Pirker. Mr. Pirker. Mr. Pirker. Ich habe für diesen Bericht gestimmt τοποθετήθηκα έτσι υπερψηφίζοντας υπέρ της ασφάλειας των παιδιών διότι ζητείται μια μεταρρύθμιση σε σχέση με πρόσθετα μέτρα για ασφαλή διαβατήρια ή βιομετρικά στοιχεία.